Εκείνη η συζήτηση ολοκληρώθηκε. Ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στι 12 το μεσημέρι. Επόμενη συνεδρίαση θα γίνει αύριο, 3η 20 Νοεμβρίου από τις ε,